Καθίστε παρακαλώ, βγάλτε τις κάρτες σας. Εισάγετε τις κάρτες σας στο μηχάνημα που έχετε μπροστά σας. πριν αρχίσουμε, θα ήθελα να καλωσορίσω μια ομάδα προσκεκλημένων της Φρανσουάς Γκροστέτ. Ε, στην ε, σημερινή ψηφοφορία είναι από την περιοχή Γον Αλπ ε, και ένα άλλο γκρουπ του Ρίχαρτ Ζίμπερ. Καλωσορίσατε όλοι. Πολύ ωραία που είσαστε εδώ και θα αρχίσουμε τώρα με την ε, ψηφοφορία αφού έχετε ετοιμάσει όλοι τις κάρτες σας. Αρχίζουμε με την έκθεση του κυρίου Ούσκη. Η των μηχανοκίνητων οχημάτων, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία παρακαλώ. Die Grünen haben einen so viel, wir müssen die Stimme von... Ε, έχουμε έναν υπεράριθμο, ο Καρλ So, jetzt können wir schließen. Λοιπόν, Εγκρίνεται 45 υπέρ, 11 κατά και μία αποχή. Συνεχίζουμε. Κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν συντομία να ευχαριστήσω τους και όδης για τη συνεργασία του σε αυτή την πολύ δύσκολη έκθεση. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω του εκπροσώπους της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Χρειάστηκε πολύ καιρό για να επιτευχθεί η συμφωνία. Αλλά πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μια εξαιρετική συμβαστική λύση. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα καταλαβαίνω γιατί κράτησε τόσο πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Συνεχίζουμε τώρα με την έκθεση της κυρίας Γκαρντίνη για το πρόγραμμα Κοπέρνικους. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, εγκρινέται 21 ε, υπέρ, κατά, αποχές, να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 21. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 7 μέρος 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 7 τμήμα 2 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 23 και 33 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά 24 άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν πολύ σαφές ας ανοίξουμε την 26 ηλεκτρονικά ξεκινάει η ψηφοφορία για την 26 ψηφανάπαντες κλείνει η ψηφοφορία σωστό 41 υπέρ 19 κατά εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές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 17 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για το ολοκείμενο άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Κλείνει ψηφοφορία. 54 υπέρ, 0 κατά, 4 αποχές. Συγχαρητήρια την... στην κυρία Συγγήτρια, την κυρία Γκαρντίνη. Θα συνεχίσουμε τώρα. Weiter geht's mit dem Bericht von Frau Antonescu. Συνεχίζουμε τώρα με την έκθεση της κυρίας Αντωνέσκου. 17 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά. Αποχές Δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 18. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν Κλείνει ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά να ελέγξουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για 19. Ψήφισαν άπαντες. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 22 υπέρ ε, άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες πέρας ψηφοφορίας για την 22 εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 και 24 μαζί υπέρ κατά εγκρίνεται 3 και 25 ίδιες υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνονται να τι ελέγξουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία για τις 3 και 25 ψηφσανάπαντες κλείνει η ψηφοφορία ε, εγκρίνονται 4 και 26 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ και 5 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 και 32 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 7 και 33 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 34 υπέρ κατά απο, απορρίπτονται 35 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 36 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 και 8 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 9 και 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 10 και 40 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά τις 10 και 40 μαζί άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 41 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ Κα... Ας ελέγξουμε τη 44 ηλεκτρονικά έρχεται ψηφοφορία για την 44 ψήψαν πάντες πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 44 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 48 υπέρ ε, συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία ψήψαν πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα περνάμε στην 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ καταπίπτει 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές ελέγχουμε τη 14 ηλεκτρονικά Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Όχι, δεν ψηφίζουμε για αυτήν. Για 16. Περνάμε λοιπόν για την καταπληκτή. Φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντε. Πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται 62 υπέρ, μία ψήφος κατά μόνο. Να ψηφίσουμε άλλη μια φορά. Άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν άπαντες. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τώρα όσον αφορά το άρθρο 70. Το θέλουμε ή όχι. Ναι. Γιατί βλέπω να γνέφουν κάποιοι. Χρειαζόμαστε 36 για ψήφο. Ψήφισαν άπαντες, άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Κλείνει η ψηφοφορία. 60 υπέρ, 3 κατά. Εύχομαι ότι καλύτερο για τις διαπραγματεύσεις. Συγχαρητήρια. So, jetzt geht's weiter im Text mit der Συνεπώς συνεχίζουμε και θα ψηφίσουμε για την εισήγηση σχετικά με το μέλι. Πρόκειται για μια εισήγηση περίπλοκη και μια ψηφοφορία περίπλοκη. Ίσως κάποια στιγμή θα χρειαστεί να διακόψουμε λίγο για να δούμε πώς θα ψηφίσουμε. Συγκεντρωθείτε αγαπητοί συνάδελφοι, θα αρχίσουμε 37, 38 και 60. Ψηφίζουμε για όλες τις τροπολογίες αυτές μαζί, κατά, Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε, ψηφίσατε όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 39 και 40 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά σχετικά με την 39 και 40. Ψήφισαν όλοι. πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε λοιπόν μετά από αυτήν την επαλήθευση με την τροπολογία 46, 46 επαναλαμβάνω, υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 46, άρχεται η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ενοποιημένο 1, ενοποιημένη 1 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συνεχίζουμε με 61-62 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 63. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 9. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 9. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με την 25 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Έλεγχος ηλεκτρονικός για την 21. Ψήφισαν όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίθηκε. Ευτυχώς που ελέγξαμε. 22 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος ηλεκτρονικός για την 22. Ψήφισαν άπαντες. πέρα τη ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 34 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 19 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Έλεγχος ηλεκτρονικός για τη 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε όντως. 36 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Ίσως θα μπορούσαμε και για μια φορά που έχουμε ήλιο, ίσως θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε τις Περσίδες. 24 υπέρ, κατά, αποχές απορρίφθηκε. Αρχίζουμε τώρα με την πρώτη τελική ε, ψηφοφορία ε, και θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι για το σχέδιο εισήγηση έτσι όπως τροποποιήθηκε. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. 47 υπέρ, 17 κατά. Ψηφίζουμε τώρα για το σχέδιο ψηφίσματος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. 47 ε, υπέρ, 13 κατά. Τώρα θα δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια, κυρία Γκέρλινγκ. Θέλετε εντολή για διαπραγματεύσεις. Αν αυτή είναι η περίπτωση, να μου πείτε ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν ζητώ εντολή, όχι. Frau Görling, Frau Görling fragt nicht um ein Mandat. Ich sehe auch keine weiteren. Κυρία Γκέρλινγκ δεν θέλει εντολή και δεν βλέπω κανέναν άλλο που θα ήθελε εντολή διαπραγμάτευσης. Συνεπώς κλείνουμε εδώ και θα συνεχίσουμε με την επόμενη εισήγηση. Περνάμε τώρα στην εισήγηση του Chris Davis. Όσοι επιθυμούν να αποχωρήσουν από την αίθουσα παρακαλώ να το κάνουν σιωπηλά προτού ψηφίσουμε για αυτήν την εισήγηση με ησυχία παρακαλώ. Αρχίζουμε. Ένα ενωπημένο υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Μετά 25. 25. 25 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε γιατί δεν είναι σαφή τα πράγματα. 25 ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα ερχόμαστε στην ενοποιημένη. 2 υπέρ, κατά, αποχές, δεν συμμετείχε. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 37 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφή τα πράγματα, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν άπαντες, πέρα στις ψηφοφορίες, εγκρίθηκε. 38 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Ενωπημένη 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. Ενωπημένη. 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε επίσης. Συνεχίζουμε με τη 45 υπέρ, κατά, αποχές δεν είναι σαφή τα πράγματα, ελέγχουμε ηλεκτρονικά για τη 45. Ψήφισαν άπαντες, Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με την ενοποιημένη 7. Υπέρ. Κατά. Οι πράσινοι έχουν την πλειοψηφία με τέσσερις ψήφους κατά. Ίσως θα πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ενοποιημένη 7. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 54 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Ενωπημένη 5 υπέρ κατά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 5 Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 36 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 63. 63 ήταν, όχι 36. Συνεχίζουμε με την ενοποιημένη 6. Κατά. Ελέγχουμε για την 6. Συμμετείχαν όλοι πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 79 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Επίσης 80 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. Επίσης 82 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 81 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 83 εισηγητού υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 84 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 85 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 86 υπέρ, κατά, απο... εγκρίθηκε, εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε, θα ελέγξουμε για την 86. Ψήφισαν άπαντες, πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. 87 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίθηκε. 88 θα ελέγξουμε για την 87 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν άπαντες, Πέρα της ψηφοφορίας, 88 υπέρ, κατά απορρίφθηκε. Ενοποιημένη 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. ...94 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε, ενοποιημένη 10, κατά, εγκρίθηκε. 97 υπέρ, κατά, Απορρίφθηκε. Ενοποιημένη 11 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 97. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν άπαντες. Πέρας της ψηφοφορίας. Χωρίς σχόλια. Ενοποιημένη 11 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. Ενωπημένη 14 υπέρ κατά εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε ενωπημένη 12 υπέρ κατά απορρίφθηκε. Θα ελέγξουμε όμως, θα ελέγξουμε γιατί τη 12, 12, 12. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν άπαντες. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 118, 119 το ίδιο υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 120 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 121 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 122 Θέλει κανείς να ελέγχουμε, ελέγξουμε για την 121. Ψήφισαν άπαντες, πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 122 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 123 και 124 μαζί υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 126 υπέρ, κατά, Απορρίφθηκε. 128 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 125 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 127. Καταπίπτει. 129. 130. Μαζί. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 132 υπέρ. Κατά. Όχι, δεν είναι σαφή τα αποτελέσματα. Ε, ελέγχομαι ηλεκτρονικά για την 132. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 133 υπέρ, κατά, Όχι, δεν είναι σαφή τα αποτελέσματα. Ελέγχομαι ηλεκτρονικά για την 133. Ψήφισαν άπαντες. Απορρίφθηκε. 138. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 135. Υπέρ. Κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 135. Ψήφισαν άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 136 υπέρ. 136 υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 136. Ψήφισαν άπαντες πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 137 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Ενωπημένη 15 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 140 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 1 υπέρ, κατά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψήφισαν άπαντες. πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 16 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 5 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 6 υπέρ κατά, απορρίφθηκε 7 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε 8 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε 9 υπέρ, κατά, ελέγχουμε ηλεκτρονικά, την 9 όλοι ψήφισαν. 9. Ψήφισαν άπαντες, πέραση της Εγκρίθηκε. 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίθηκε. 11 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. 9 υπέρ. Κατά εγκρίθηκε. 13 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 14 υπέρ κατά απορριφθήκε. 15 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 16 υπέρ κατά εγκρίθηκε. αιτιολογική ε, σκέψη ήτρε σε απορριφθήκε. Δι υπέρ. Α, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη ΣΥ ήτρε. Ψήφισαν άπαντες πέρα της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Δε ήτρε υπέρ κατά απορρίφθηκε. Ε, ήτρε υπέρ κατά απορρίφθηκε. Παράγραφος 2 Ήτρε υπέρ κατά εγκρίθηκε. Ενωπημένη 17 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 6 υπέρ κατά εγκρίθηκε. 8 υπέρ κατά απορρίφθηκε. 9 υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 10 υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. 11 υπέρ. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 10. Ψήφισαν όλοι. Απορρίφθηκε. 11 ήτρε υπέρ, κατά Απορρίφθηκε. 16 ήτρε. Υπέρ, κατά, εγκρίθηκε. 18 ήτρε. Υπέρ, κατά, απορρίφθηκε. Α, εγκρίθηκε. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρα τη ψηφοφορίες, εγκρίθηκε. 20 ήτρε υπέρ κατά απορρίφθηκε. Και τώρα ερχόμαστε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Όλοι ψήφισαν πέρα στις ψηφοφορίες. 51 υπέρ 2 κατά μία αποχή εγκρίθηκε ε, συγχαρητήρια στον Κρίς Ντέιβις. Θέλετε να ζητήσετε εντολή. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κοιόδης εισηγητές που με τη συμβολή τους βοήθησαν στην ενοποίηση των τροπολογιών που βελτίωσε σημαντικά την αρχική μου έκθεση και τώρα έχουμε μια σαφή δήλωση προς την Κομισιόν που θα παρουσιάσει κάποιε ωραίε ιδέε που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτή τη τεχνολογία που έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση των ε, ανθρακούχων εκπομπών στην ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Κρυστέιβι. Προχωράμε με την έκθεση του συναδέλφου Βιτόριο Πρόντι. Και αρχίζουμε ευθύ αμέσω με την συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα, προχωράμε στην 55, υπέρ. Κατά. Γιατί δεν συμμετέχουν οι σοσιαλιστές. Βαριέστε. Η κυρία Κοντμπέρεντ λέει πως βαριέστε. Λοιπόν, 55 ξανά, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προχωράμε με το 4α, έτσι για να μην βαριέστε κιόλα, ενοποιημένη υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση αμέσως της 4α. 4α εννοποιημένη. Σελίδα 7. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνατε. Καταπίπτει λοιπόν 4β και περνάμε στην 148, 10 σελίδα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 148. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προχωράμε. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά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 Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 1. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλη 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεν ψηφίζουμε την 9, περνάμε στην συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 ερτούγκ υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατά τμήματα 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία, όπως πάντα ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε. Πέρας. 60 θετικές ψήφοι, μία αρνητική, εγκρίνεται, συγχαρητήρια στο Βιτόριο Πρόντι. Βιτόριο, παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη στήριξή τους και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη βοήθεια που έλαβα από το προσωπικό μου τον ε, Δ. Σαγκράσο. Ήταν πολύ δύσκολη η εργασία μας ε, για να καταφέρουμε να ε, διατυπώσουμε σωστά τις συμβιβαστικές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην έκθεση της Πιλάρα σου. Αρχίζουμε. Ίνκο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την Φεμ 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Φέμε νέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μόνο ένα συμμετείχε στην ψηφοφορία. Οι υπόλοιποι που είστε. Ξανά ψηφίζουμε. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Άρα λοιπόν καταπίπτουν οι υπόλοιπε τροπολογίε της ΦΕΜ. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σελίδα 3. ανα. Πάμε στην συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έτσι για να μην βαριόμαστε κιόλα. Φέμ 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι η ηλεκτρονική επαλήθευση. ΦΕΜ 18 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. ΦΕΜ 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 74 τέσσερα υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 74. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 11. Όχι, καταπίπτει. Ήμκο 11. 76. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρο, καταπίπτει και αυτή. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα τη τροπολογία 76. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Φεμ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ, απορρίπτεται. Φεμ 3. Υπέρ. Κατά. αποχέ, απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ίνκο 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Α νέα υπέρ κατά Α, μάλιστα. Όχι, πάμε στη ΦΕΜ 1, διορθώνω. ΦΕΜ 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 97, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 101, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99 και μέχρι 100 ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 109 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ενοποιημένη β υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 3 υπέρ, κατά αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την ΙΝΚΟ 3. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 ή κατά πίπτη 121 122 λοιπόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ίνκο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 κατά πίπτη, φεμ 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Φεμ 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμικο 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 κατά πίπτη και πάμε στην Ήμικο 12. Όχι κατά αυτή. Άρα πάμε στην φεμ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φεμ 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φεμ 14 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φεμ 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέγγι 3. Καταπίπτει η Ρέγγι 3 και πάμε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 Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 και ενωπημένη 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έτσι. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Ενοποιημένη α. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Και 51 υπέρ, κατά, αποχές, δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 51. Ψηφίσατε. Πέρας. Μάλιστα, απορρίπτεται, σαφέστατα. Περνάμε τώρα στην ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. «62 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή, συγχαρητήρια». weiter geht's. Συνεχίζουμε με την έκθεση Έστερ Δελάνια. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε. Αρχίζουμε λοιπόν. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Όχι, δεν είναι σαφές, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 43. Ψηφίσατε. Πέρας. 27 θετικές, 33 αρνητικές απορρίπτεται. Ενοποιημένη 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 49. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άγκρι 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κάποιος μιλάει ή στο τηλέφωνο με το διπλανό του. Δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά ενοχλεί. Ευχαριστώ πολύ. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Πέρας. Απορρίπτεται. 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 75. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Άποχες. Απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 80. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Άγκρι 16 και την άγκρι 6 δεν τις ψηφίζουμε. Πάμε στην 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 87. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίφθηκε. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνατε. 92 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνατε. 94 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση πρώτο τμήμα της 94. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 για την τροπολογία 98 υπέρ με την προφορική τροπολογία. Κατά. Εγκρίνεται. Άρα περνάμε στην ενοποιημένη 7. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 107. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ούτε εδώ είναι σαφές. Ψηφίζουμε και την 101 ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114 υπέρ. Όχι, θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 113, μιας και το ζητήσατε. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε, πέρασε. Εγκρίνεται. 114. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 116. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Καταπίπτει. 121 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Άγκρι 7. Δεν την ψηφίζουμε. Προχωράμε στην άγκρι 14. Όχι, ούτε αυτή ψηφίζουμε. Άρα, τροπολογία 124 χωρίς του Σνέλχαρτ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ήμκο 8. Υπέρ. Όχι, καταπίπτει Ίμκο 8 και η επόμενη και περνάμε στην 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 131 με προφορική τροπολογία. Πρώτο τμήμα α υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα, 135 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 136, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 137, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 137. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 140 καταπίπτει, 141. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άγκρι 15. Υπέρ. Κατά.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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Την ψηφίζουμε, ναι. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές. Ηλεκτρονική επαλήθευση 24. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ενοποιημένη 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές... Όχι καταπίπτει. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Καταπίπτει 36, 37. Υπέρ. Κατά.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 42 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Όχι. Με συγχωρείτε, δεν ήταν σαφές. Θα επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά και την 42. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Συγχαρητήρια, Έστερ ομόφωνα 58 ψήφοι υπέρ. So, jetzt haben wir... Μάλιστα, εγκληματικό τρισβάρος άγριων ειδών τώρα.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 Όχι, με συγχωρείτε, ήταν και οι δύο μαζί. Πάμε στη 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 38. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ. Κα... 47. Μου λέτε και αποκεκτημένη ταχύτητα. Όχι. Θέλετε να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά τη 42. Μου το ζητάτε, το απαιτείτε. Ορίστε, πάρτε το. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 7 47 υπέρ. Κατά. Αποχές θα κοιτάξουμε η ηλεκτρονική επαλήθευση. Για την 47. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 43 αποσύρθηκε. 44 και 45 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεν είναι σαφές. Η ηλεκτρονική επαλήθευση Γιατί τις 44 και 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Πέρας. Εγκρίνονται. 49. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 51. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές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 70 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 73 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, δεν είναι σαφές η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 78. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. η Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 82. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα το συζητήσουμε και στο μέλλον αυτό. 83. Υπέρ. Κατά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 Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 57 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στους εισηγητές. Και με αυτό ολοκληρώνεται η σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα συναντηθούμε με τους συντονιστές στις 9 και με τους υπόλοιπους από εσάς και με την Κόνη Χέντεγκαρτ στις 10. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο.